Αγαπητοί φίλοι, παρακαλώ. Θέλουμε να προλάβουμε να πάμε στην Ολομέλεια για να ακούσουμε τον Καναδό Πρωθυπουργό. Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί στη χρήση του χρόνου μας. Καταρχήν, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ που είστε παρόντες. Ξέρετε ότι Είχαμε λίγο χρόνο για τη συζήτηση της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων και γι' αυτό προβλέψαμε σήμερα αυτή την έκτακτη συνεδρίαση ώστε να έχουμε μια συζήτηση και οι συγγήτρια και οι συγγήτρες και οι σκιώδεις συγγητές να συζητήσουμε τους ευρωβουλευτές πολύ πιο αποτελεσματικά και με επάρκεια. Έχουμε 20 γλώσσες ε, για διερμηνία. Δεν έχουμε φιλανδικά, μαλτέζικα και γοεδελικά. Σχεδόν πλήρας καθεστώς διερμηνίας δηλαδή. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στις συγκεκριές μας. Τέσσερα λεπτά στην καθεμία. Αποφασίστε μεταξύ σας ποια θα ξεκινήσει. Η κυρία Μωράν Σαρτιά, ξεκινήστε εσείς και μετά η Άνιας Γιονγκέριους. Και μετά δύο λεπτά οι υπόλοιποι βουλευτές. Σας ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε που μας δώσετε από τέσσερα λεπτά στην κάθε εισηγήτρια. Εγώ θα το εξαντλήσω το τετράλεπτο γιατί ήδη την περασμένη φορά ήδη κάναμε μια παρουσίαση της έκθεσης, οπότε σε αυτή τη συνεδρίαση θα ήθελα να αφιερώσουμε όλο το χρόνο ε, στα σχόλια των ε, συναδέλφων που θα μας πούν ποια σημεία είναι για τις πολιτικές τους ομάδες τα πιο σημαντικά. Αυτό το κείμενο είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλες τις πολιτικές ομάδες, γιατί το κείμενο αυτό είναι σημαντικό για ολόκληρη την Ευρώπη. Θα θέσουμε με το κείμενο αυτό τα θεμέλια της κοινωνικής Ευρώπης. Γι' αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε σήμερα σε αυτό το θέμα και κυρίως στα πιο σημαντικά ζητήματα της αμοιβή των αποδοχών, ε, της διάρκειας, της νομικής βάσης, των γραφείων μερικής απασχόλησης ε, και της απόσπασης ε, εδώ Αυτά και περιμένω τα σχόλια των συναδέλφων, γι' αυτό δεν θα εξαντλήσω το χρόνο μου. Ούτε κι εγώ χρειάζομαι το δίλεπτο. Να ευχαριστήσω απλώ του συναδέλφου που ήρθαν για να συζητήσουμε σήμερα γιατί ξέρω ότι όταν προγραμματίζουμε έκτακτες συνεδριάσεις είναι δύσκολο να ε, είμαστε παρόντες. Αλλά χρειάστηκε αυτή η έκτακτη συνεδρίαση γιατί δεν προλάβαμε την περασμένη φορά να ολοκληρώσουμε μια ευρεία και ανοιχτή συζήτηση για το θέμα αυτό της απόσπασης των εργαζομένων. Γι' αυτό σήμερα την πρωινή μας συνεδρίαση θα ήθελα να την αφιερώσουμε ολόκληρη στη συζήτηση, να ακούσουμε τις απόψεις των Ευρωβουλευτών. Στόχος μας είναι να καταλήξουμε σε μια ισορροπημένη ε, έκθεση που θα συγκεντρώσει όσο το δυνατό μεγαλύτερη πλειοψηφία και στην Επιτροπή και κατόπιν και στην Ολομέλεια. Γι' αυτό θέλουμε να ακούσουμε όλους τους συναδέλφους, να αφουγκραστούμε τις ανάγκες τους. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Περιμένω τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Χότς που εκπροσωπεί τους φιλελευθέρους είναι παρόν. Ή μάλλον όχι από τις μεταρρυθμιστές συντηρητικού. Όχι, κυρία δεν πάλω από τους φιλελεύθερους τώρα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δύο λεπτά είπα στον καθένα. Ευχαριστώ. Διάβασα προσεκτικά την έκθεση και θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ε, δύο συνεισηγήτριες, γιατί πραγματικά βρήκαν μια σωστή ισορροπία μεταξύ τους. Βέβαια, δεν είναι μυστικό ότι ε, δεν είμαι ενθουσιώδης υπέρμαχος πρότασης ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα καταθέσω τραπολογίες για μερικές αλλαγές, αλλά θεωρώ ούτως ή άλλως ότι η προτινόμενη αναθεώρηση ήταν περίτη, γιατί συνεχίζονται ακόμη οι μεταθέσεις των εκτελεστικών οδηγιών. Πάντως θεωρώ ότι η ελεύθερη διακίνηση των προσώπων και των υπηρεσιών είναι σημαντική, για να μην πω η σημαντικότερη ευρωπαϊκή αξία. Εδώ μιλούμε για την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών. Θεωρώ ότι η διαφορετικότητα και η πολυμορφία στην Ευρώπη είναι απαραίτητη προπόθεση για την ανταγωνιστικότητα. Και φέτο έμαθα να ακούω και την άλλη γνώμη, ε, να ακούω την κοινή γνώμη ε, των χωρών που επίμονα ζητούσαν αυτή την αναθεώρηση και τώρα άρχισα να καταλαβαίνω, να αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες αυτών των χωρών αλλά θα ήθελα να ζητήσω αντίστοιχη κατανόηση και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή θα ήθελα και οι χώρες που ζητούν την αναθεώρηση να ε, κατανοήσουν τις ανησυχίες και τους ενδιασμούς των χωρών που είναι κατά της αναθεώρησης. Φυσικά θέλουμε να διευκολύνουμε την ε, παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών και να βελτιώσουμε τη λειτουργία της ε, εσωτερικής αγοράς και φυσικά θα πρέπει να είναι ε, ευανάγνωστο το κείμενο και εύχριστο, αλλά έχω τρία συγκεκριμένα θέματα. Καταρχήν, την εφαρμογή της πρότασης σε όλους τους τομείς. Με προβληματίζει το γεγονός ότι καλύπτονται όλοι οι κλάδοι από την πρόταση αυτή, δηλαδή και οι μεταφορές και οι ενδοεπιχειρησιακές αποσπάσεις. Κάτι άλλο που ε, δεν έχει διευκρινιστεί είναι ο ορισμό των αποδοχών τη αμοιβή. Και αυτή η ασάφεια είναι μεγάλο πρόβλημα της πρόταση, γιατί ακόμη περιμένουμε την εξήγηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για αυτή την ασάφεια. Και θα ήθελα να ζητήσω διαφάνεια. Όλα τα στοιχεία ε, της σύνθεση των αποδοχών θα πρέπει να είναι δημόσια. Να μην υπάρχουν αδιαφάνεια τέτοια στοιχεία. Επίσης, ο κανόνα των 24 μενών δεν έχω πιστεί ότι θα λύσει το πρόβλημα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτά, για κατά τη γνώμη μου, είναι τα τρία βασικά στοιχεία που με προβληματίζουν. Έχω και άλλα, θα μπορούσαμε να συζητάμε όλες ολόκληρες, αλλά θα καταθέσω και τροπολογίες και φυσικά θα σας κρατώ ενημέρους. Δύο λεπτά και στη Ρίνα Ρόνια Κάρη από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τις συγγήτριες ε, και να τις συγχαρώ για τη μέχρι τώρα συνεργασία που είχαμε. Είχαμε πολλές συνεδριάσεις, ε, εκτενείς διαβουλεύσεις και ακούσαμε την άποψη πολλών ενδιαφερομένων. Διαβάζοντας ε, την, το σχέδιο έκθεσης, διαπιστώνω ότι έλεξαν υπόψη πολλές απόψεις και ευελπιστώ ότι θα καταλήξουμε σε συμβαστικές προτάσεις για πολλά θέματα. Ποιες είναι οι σημαντικότερες πρωτοβουλίες μας τώρα για τη συνέχεια. Καταρχήν είναι προφανές ότι θα πρέπει να ορίσουμε την έννοια της απο... των αποδοχών, της αμοιβή. Θα πρέπει να είναι σαφής αυτή η έννοια. Και φυσικά να προσδιορίσουμε ότι τα κράτη-μέλη ε, έχουν το δικαίωμα να μπορούν να προσδιορίζουν αυτή την έννοια. Και συμφωνώ ότι θα μπορούσαμε να διευρύνουμε τη συζήτηση για να καλύπτει και τις ε, συλλογικές συμβάσεις και κυρίως ε, θα πρέπει για ίση εργασία να ισχύουν και ίσες αμοιβέ σε τοπικό και κλαδικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια, να είναι προσωρινή. Η πρόταση της ΓΚΟΕ ζητά μείωση αυτής της προθεσμίας. 24 ε, μήνες είναι υπερβολικά παρατεταμένη περίοδος. Προτείνουμε εξάμεινο για να τονίζουμε ότι η απόσπαση είναι προσωρινό μέτρο. Επίσης, τελευταίο σημείο, κάτι που ήδη αναφέρατε, συμφωνώ και συμφωνούμε όλοι νομίζω ότι θα πρέπει να περιλάβουμε και ένα κοινωνικό κεφάλαιο στην πρόταση και να προσδιορίσουμε, να επισημάνουμε ότι πρόκειται για μια οδηγία ελάχιστων προϋποθέσεων και τα κράτη-μέλη, αν το επιθυμούν, μπορεί να είναι πολύ πιο φιλόδοξα. Να είμαστε σαφείς. Διεύρυνση λοιπόν της νομικής βάσης είναι απαραίτητο στοιχείο. Πάντως, όπως είπα, θα καταθέσουμε πολλές τροπολογίες, αλλά θεωρώ ότι ο διάλογος μέχρι τώρα ήταν καλός, κάτι που ε, αναγγέλει και ένα καλό μέλλον στη συνεργασία. Η Τέρι Ρέιτ και από τους Πρασίνους. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τις δύο συνεισηγήτρες και τους Κιώδης για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ε, περίοδο που περάσαμε μαζί. Θέλω να κάνω δύο γενικού φύση παρατηρήσει πριν μπω στι τροπολογίε. Η πρώτη είναι ότι υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι αν ότι αν ξεφορτωθούμε τελείω αυτή την οδηγία θα βελτίωνε την κατάσταση των εργαζομένων στην Ευρώπη. Εγώ πρέπει να δηλώσω ότι αυτό είναι ανοησία, γιατί αν ξεφορτωθούμε την οδηγία αυτή εντελώ, αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα γίνει ένα αγώνα προ τα κάτω και ότι η ελάχιστη προστασία που έχουν αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι θα ε, ε, εξαλειφθεί εντελώ. Πρέπει να είμαστε έντιμοι απέναντι στον κόσμο ότι θα υπάρχει λιγότερε ρυθμίσει θα υπάρχουν. Και αν ε, δεν ισχύσει αυτή η οδηγία, θα βγουν από την ενιαία αγορά και αυτό δεν είναι επιλογή καν για τους εργαζόμενους της Ένωσης. Και κάτι ακόμα που θέλω να πω είναι ότι συχνά στη συζήτηση αυτό που έγινε ήταν ότι ε, αυτή η οδηγία παρατίθεται στην άλλη για την επιβολή δεν θα πρέπει να αντιπαραθέτουμε αυτές τις δύο οδηγίες, γιατί χρειάζεται να ασκήσουμε πίεση σε όλα τα κρατημέλη, ώστε να μεταγράψουν την οδηγία περί της επιβολής, μόλις θα έχει ολοκληρωθεί ε, τούτη εδώ. Και μάλιστα θα πρέπει ακόμα περισσότερο να επιμείνουμε, ώστε να τα θέσουν σε εφαρμογή τα κρατημέλη. Αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε ποια είναι τα προβλήματα εκείνης της οδηγίας και γι' αυτό χρειάζεται και αυτή εδώ η διάταξη. Και τελευταία παρατήρηση που θέλω να κάνω. Οι περισσότεροι από εμά πιστεύω ότι συμφωνούμε πως θέλουμε να ε, προστατεύσουμε την ελευθερία κυκλοφορίας και υπηρεσιών. Όμως πρέπει να διερωτηθούμε ότι αν δεν υπάρχει ισότιμο πεδίο στα διάφορα κράτη-μέλη, θα γίνει αυτός ο αγώνας προς τα κάτω. Γι' αυτό χρειάζεται να αναθεωρηθεί αυτή η οδηγία για να δημιουργηθεί ένα ισότιμο πεδίο για όλους τους εργαζόμενους της Ένωσης. Τώρα, για να μπω λίγο εις βάθος στο θέμα τα που μας απασχολούν σήμερα. Ένα από τα πολύ σημαντικά είναι η νομική βάση, γιατί αυτό που έχουμε τώρα στρέφεται προς την ελευθερία των υπηρεσιών περισσότερο και δεν εξετάζει τόσο τα δικαιώματα των εργαζόμενων, που εμείς κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να είναι το πιο κρίσιμο. Δέκα δευτερόλεπτα ακόμα η ανάγκη για συλλογικές διαπραγματεύσεις, να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας στις πιο αντιπροσωπευτικές συλλογικές διαπραγματεύσεις. Είναι πολιτική φύση αυτή η συζήτηση. Φυσικά θα πρέπει να συζητήσουμε τα τεχνικά στοιχεία, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε μάλλον δεν θα πρέπει να αποσυρθούμε από αυτή τη συζήτηση λόγω και μόνο των ε, τεχνικών δυσκολιών. Ευχαριστώ. Ε, Λάουρα Αουτζέα που από το FTD δεν είναι εδώ. Ο κύριος Χόκ τώρα, ε, εξ της ΣΑΛΔΕ. Όχι, ΣΙΑΡ. Δύο λεπτά έχετε. Είμαι ικανοποιημένος που έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων σήμερα. Πριν να καταθέσουμε αυτές τις τροπολογίες και να αρχίσουμε τη συζήτηση και την εργασία σε αυτή την πρόταση, επ' αυτής της πρότασης, είναι σημαντικό εμείς ως αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής θα πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι τα διακυβεύματα. Θα πρέπει να αποφύγουμε το διχασμό της Ευρώπης ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση η πρόταση αυτή δεν θα πρέπει να αφορά ε, μια τέτοια διαίρεση. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε που υπάρχουν τα βασικά προβλήματα και να βρούμε ρεαλιστικές και λειτουργικές λύσεις για τα κράτη-μέλη και τους εργαζόμενους τους και τις επιχειρήσεις τους. Θα ήθελα να παροτρύνω τους συναδέλφους να εξετάσουν αυτή την πρόταση ως έναν τρόπο για την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Πρέπει η πρόταση αυτή που αφορά τους αποσπασμένους εργαζόμενους να λειτουργήσει τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις. Συμφωνώ ότι πρέπει να καταργηθούν τα παραθυράκια που μπορεί να διευκολύνουν τις αποσπάσεις Αλλά δεν μπορούμε να λύσουμε το θέμα το γενικότερο της εκμετάλλευσης των εργαζομένων με αυτήν εδώ την οδηγία. Χωρίς να μπω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες σήμερα εδώ, υπάρχει ένα θέμα κλειδί που θα ήθελα να αναφέρω. Όταν μιλάμε για επιχειρησιακές ε, μετακινήσεις, αποσπάσεις εργαζομένων, είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε ότι δεν αναφερόμαστε μόνο σε εργαζόμενους στον κατασκευαστικό τομέα, αλλά μιλάμε και για τεχνικούς επαγγελματίε, αλλά και για ε, πτυχιούχους που κινούνται από τη μια χώρα στην άλλη, ενώ εργάζονται για την ίδια εταιρεία. Moment. Ε,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 η γνωμοδότηση αυτή πιστεύω πως ε, είναι πραγματική πρόκληση και προσβολή απέναντι σε αυτές τις δύο κυρίες που εργάζονται εδώ και έξι μήνες. Γνωρίζοντα ότι στην τελευταία επιτροπή, λόγω δικού σα φάλματος, γιατί κυρία Πρόεδρε δεν ελέγχεται ούτε τα ωράρια ούτε τους χρόνους ομιλίας, αναβλήθηκε αυτή η επιτροπή συνεδρίαση. Και ανανεώνω λοιπόν τη συγνώμη εκ μέρους μου και εκ μέρους σας στις δύο γιατί αυτό που κάνετε είναι απαράδεκτο για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Για να δώσω τώρα τη θέση μας. Ε, το πρώτο σας ε, λεπτό το χρησιμοποιήσατε για να διαμαρτυρηθείτε. Κυρία Πρόεδρε, η υπεροψία σας φτάνει πια. Μόνο και μόνο απέναντι στι συνεισηγήτρε θα έπρεπε να δείχνετε καλύτερο, περισσότερο σεβασμό. Όσο και αν βάζετε το καλό σα χαμόγελο, είστε απαράδεκτοι. Κύριε Κάζα, κύριε Κάζα, ο κύριος Κάζα δεν ακούγεται, είναι χωρίς το μικρόφωνο. Κύριε Πρόεδρε, Δεν μπορώ να δεχτώ αυτά τα λόγια από έναν συνάδελφο. Όλοι συμφωνήσαμε πως θα έχουμε τον ίδιο χρόνο. Είτε είσαι από το ΕΛΚ, το ΑΛΔΕ, το ΙΕΝΕΦ ή οπουδήποτε, θα πρέπει να ε, ε, συμπεριφέρεσαι με τον ίδιο τρόπο και να... Κύριε Ντομινίκ Μαρτά, σταματήστε και, και, και πείτε μας την ερώτησή σας. Κύριε Μαρτά, τέλειωσε ο χρόνος σας. Προχωράμε στον εκπρόσωπο της Γιούρη εκπρόσωπο για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γιούρη. Ε, ε, ε, οι εξαλλοσύνες σας αυτές δεν σας εξυπηρετούν. Η λαϊκίστικη αυτή συμπεριφορά σας φαίνεται γιατί μαγνητοσκοπείτε και θα βγει έξω από εδώ. Και κύριε Κάζα, το τουπέ σας φτάνει. Κύριε Μαρτέ, μη μας κάνετε να χάνουμε το χρόνο μας. Έχουμε σοβαρή δουλειά εδώ μέσα. Ναι, μα εγώ αντιπροσωπεύω εκατομμύρια εκλογή. Αυτό σα εξοργίζει ότι έχω τόσα εκατομμύρια πίσω μου. Ναι, ναι, αλλά σας ευχαριστώ γιατί αυτά όλα μαγνητοσκοπούνται και θα βγουν έξω από αυτή την αίθουσα, θα βγουν στις τηλεοράσεις. Thank you. I will now give the floor. Yes, please, please. Uh, ναι, επειδή ακριβώς καταγράφονται όλα αυτά, θέλω να πω ότι ο, η πριν, ο ομιλητής πριν από τον κύριο Μαρτέ δεν αντιπροσώπευε την Άλντε, γιατί δημιουργήσατε μια σύγχυση. Είπατε ότι είναι μέλος της Άλντε και θέλω να το υπογραμμίσω, δεν είναι της Άλντε. Ναι, η, η πρόεδρος είπε πρώτα, τον παρουσίασε, πως ήταν από την Άλντε. Ναι, το διόρθωσα. Λοιπόν, ο κύριος Ρολάου ζήτησε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι σε ένα τέτοιο θέμα, για να διορθώσουμε πολλά προβλήματα, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η έννοια της απόσπασης. Τι θα πει απόσπαση. Η απόσπαση είναι κάτι που επιτρέπει σε επιχειρήσεις που που επιτρέπει σε, επιχειρήσεις που έχει δραστηριότητα σε μια άλλη χώρα να αποσπάσει για, για κάποια περίοδο τους εργαζομένους της στην άλλη χώρα. Οπότε το βασικό πρόβλημα αφορά κάποιες πρακτικές που δεν ανταποκρίνονται σε αυτή τη φιλοσοφία. Δηλαδή, η ταγραφία μερικής απασχόλησης, ε, η ψευτοαπασχολούμενη ή αυτοαπασχολούμενη ή η συσσόρευση ε, εργασιών θα πρέπει να διευκολύνουμε υπεργολαβιών. Ε, θα πρέπει να αποφύγουμε τον ε, ανταγωνισμό μεταξύ των εργαζομένων μόνο και μόνο για να ρίξουμε το κόστος. Και με βάση αυτή τη φιλοσοφία μπορούμε να χαράξουμε μία γραμμή και να διαχωρίσουμε τα ενδιαφέροντα σημεία από αυτά που είναι περιτά. Επίσης, ε, σε ό,τι αφορά την έννοια της αμοιβή των αποδοχών, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να σεβαστούμε και τις εργασιακές και τις βιωτικές συνθήκες των αποσπασμένων εργαζομένων. Για παράδειγμα, στη χώρα μου ε, γίνεται απόσπαση εργαζομένων και ο εργοδότης σέβεται την νομοθεσία που λέει ότι αν δεν πληρώσει αποζημίωση για τη στέγαση θα πρέπει να εξασφαλίζει στέγαση και συνήθως τους βάζουν σε εμπαρευματοκιβώτια για να στεγάζουν αυτούς τους εργαζομένους που τους έχουν αποσπάσει. Αυτό όμως είναι παράδεκτο. Σας ευχαριστώ. Και τώρα να δώσω το λόγο στον Εμίλιο Πάφ. Ναι, είστε άξιος εκπρόσωπος της ε, ακροδεξιάς και γνωστός αντιευρωπαίος. Δυστυχώς εκτός σχολείου τα σχόλια του κύριου Μαρτά. Αν θέλετε να μας δίνετε έξω από την αίθουσα να το κανονίσουμε. Ο λόγο στον κύριο Πάβελ. Επειδή έχουμε λίγο χρόνο, ευχαριστώ κύριε Μαρτάμπ. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι μα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνουμε μάχη για καλύτερη προστασία των εργασιακών συνθηκών όλων των Ευρωπαίων εργαζομένων από όπου και αν προέρχονται ε, και σε όποια χώρα και αν είναι απαραίτητε οι υπηρεσίε του. Και εγώ σέβομαι την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών και εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά φοβάμαι ότι κάνουμε κακό παρακαλώ, γιατί με την υπερβολική ρυθμίση ε, δυσκολεύουμε αυτούς τους νομοταγείς ε, εργοδότε και εργαζομένους. Δεν θέλουν να διαλέγουν οι επιχειρήσεις μεταξύ του να κλείσουν ή να ε, μετακινηθούν στην αδήλωτη εργασία. Δεν θέλω επίση οι αποσπασμένοι να μετατραπούν σε μόνιμα εργαζομένου ή να κερδίζουν περισσότερο από ότι οι συνάδελφοί τους στην πατρίδα τους. Αυτό είναι παράδοξο. Θέλω ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών ε, υπηρεσιών και εργαζομένων, χωρίς όμως να ορθώνουμε περισσότερα εμπόδια από αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε, για παράδειγμα, στο Σέγγεν. Επίσης, έχουμε μια καλή οδηγία για την εφαρμογή. Πολύ φοβάμαι ότι η νέα οδηγία για την απόσπαση θα αποτύχει στην υλοποίηση των δηλωμένων στόχων της και θα ωφελήσει μόνο ένα πολύ μικρό αριθμό εργαζομένων οι, η αποσπασμένοι ε, που υποτίθεται, υποτίθεται εργαζομένοι που ζουν στο δρόμο δεν θα πρέπει να είναι αντικείμενο της ε, συζήτησης αυτής. Θα πρέπει ε, να αντιμετωπίσουμε το πραγματικό πρόβλημα κατεπηγόντως άσχετα με τις εθνικές πολιτικές και, δράσεις και τις προεκλογικές εξτρατείες που έχουμε φέτος. Θα πρέπει να χτυπήσουμε τις αδήλωτες πρακτικές όπως το δουλεμπόριο, ή της, την ψεύτο αυτοαπασχόληση. Θα πρέπει επίσης να στηριζόμαστε σε πραγματικά περιστατικά και να μην α, συγχαίουμε τις αθέμητες και παράνομες πρακτικές με το θέμα της απόσπασης. Να προστατεύσουμε εκατομμύρια Ευρωπαίους από εκμετάλλευση, εξαθλίωση και από αβέβαιο και σκοτεινό μέλλον. Και η ιδέα ότι η απόσπαση από λιγότερο εύπορες χώρες σε πιο εύπορες ε, είναι κοινωνικό ντάμπινγκ ε, είναι λάθος γιατί ακόμη και χώρες από πιο ανεπτυγμένες ε, επιχειρήσεις από πιο ανεπτυγμένες χώρες επενδύουν ακριβώς σε λιγότερο ανεπτυγμένες ακριβώς λόγω του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που τους δίνει το χαμηλό εργασιακό κόστος. Μήπως αφιβάλλεται ότι και αυτοί οι άνθρωποι θα ήθελαν να έχουν καλύτερους μισθούς στις πατρίδες τους. Ευχαριστώ κυρία Κοζουόφσκα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ο στόχος της οδηγίας είναι η προστασία των εργαζομένων, των δικαιωμάτων των εργαζομένων και η αύξηση της διαφάνειας των διατάξεων, διευκολύνοντας τις αποσπάσεις για τις επιχειρήσεις. Ε, οι εμπειρογνώμονες ε, μας διαβεβαίωσαν ε, ότι με την οδηγία αυτή θα επιβαρύνουμε το έργο των επιχειρήσεων και θα δημιουργήσουμε πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιλύουμε, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχω την αίσθηση ότι με την πρόταση αυτή θα υποφεληθούν οι μεγάλες επιχειρήσεις, κυρίως της Δυτικής Ευρώπης, και θα βγουν χαμένες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως της Ανατολικής Ευρώπης. Για παράδειγμα, οι μεταφορικές εταιρείες, που καλύπτονται από άλλη οδηγία. Εδώ δεν έχουμε ειδικέ ε, ε, διατάξει για τι μεταφορέ. οπότε ό,τι μα λείπει από την οδηγία αυτή δεν θα ισχύει για τι μεταφορέ, Ενώ 80% των επιχειρήσεων του κλάδου των μεταφορών είναι μικρομεσαίες επιχειρήσει, κυρίω μικρέ επιχειρήσει που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτή την τεράστια γραφειοκρατική επιβάρηση που επιφέρει αυτή η πρόταση. Επίσης, για την αμοιβή. Δεν είναι γνωστό το θέμα της αμοιβή, ούτε οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν το γεγονός ότι αν ε, με τις μεταφορές ε, ο οδηγός περνάει από πολλές χώρες ε, τι ισχύει για κάθε, σε κάθε χώρα αυτή, σε κάθε από τις χώρες αυτές για την αμοιβή. γιατί κάθε χώρα έχει τη δική της γλώσσα και θα πρέπει η μικρή επιχείρηση να γνωρίζει όλες αυτές τις διατάξεις στις ενδιάμενες χώρες. Στην ε, Πολωνία, για παράδειγμα, έχουμε το εξή παράδειγμα. Αν ο οδηγό περνάει για 90 μέρε διάφορε χώρε, ε, από η διαφορά μπορεί να είναι μέχρι και 1500 ε, ευρώ, ανάλογα με το, το ποιε χώρε περνάει. Οπότε, ποια είναι η ισότητα μεταξύ των εργαζομένων. Υπάρχει μια σωρία προβλημάτων που δεν τα λαμβάνουμε υπόψη στην οδηγία αυτή. Όλα αυτά θα πρέπει να τα εξετάσουμε και γι' αυτό θα καταθέσω και τροπολογίες στην έκθεση. The Lenners, two minutes. Ευχαριστώ, Λέναρ, σε δύο λεπτά. Um, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Τελικά το σημερινό πρωινό πολύ ενδιαφέρον και είμαι χαρούμενος που θα γυρίσω στην Ολλανδία και θα μπορέσω να εξηγήσω ότι οι συνέδελφοι από το Εθνικό Μέτωπο ε, φωνάζουν, ε, λένε, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα θέματα που ασχολούν τους ε, ψηφοφόρους και τα θέματα υπάρχουν και όσον αφορά την απόσπαση των εργαζομένων. Εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε για την ελεύθερη μετακίνηση, διακίνηση των υπηρεσιών, όχι μόνο μετακίνηση των εργαζομένων που είμαι υπέρ. Όλοι οι εργαζόμενοι σε όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε θα πρέπει να είναι ελεύθεροι και είναι ελεύθεροι να εργαστούν σε οποιαδήποτε χώρα επιτιμούν. Με, τις, με τους ίδιους όρους όπως και οι ντόπιοι εργαζόμενοι. Αλλά πολλέ φορέ η απόσπαση εργαζομένων χρησιμοποιείται ω ένα τέχνασμα για να παρακάμψει κανεί αυτή την ελεύθερη μετακίνηση εργαζομένων. Νομίζω ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για τη διάρκεια της απόσπαση Λέμε ότι για μικρό χρονικό διάστημα. Μα πόσο δεν το ορίζουμε αυτό, πρέπει να το ορίσουμε. Οι πολιτικοί πρέπει να πούν τι κατά την άποψή τους, ε, πότε κατά την άποψή τους ή για πόσο χρονικό διάστημα μπορούν να αποσπούνται οι εργαζόμενοι. Ε, μερικοί πιστεύουν ότι θα πρέπει να είναι μικρότερο το διάστημα από άλλους, άρα δηλαδή θα πρέπει να βρούμε καινοτόμους τρόπους για να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Και συμφωνώ απόλυτα με την Ελισαπέτα και τον Άχνες ε, και την Άγνες, με συγχωρείτε, για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα. Ε, αυτή τη στιγμή είναι απαράδεκτο οι αποσπαζόμενοι να εργάζονται μαζί με τους ε, γηγενείς, οι οποίοι εργάζονται με ακατάστατους όρους ε, και οι αποσπασμένοι όχι. εργάζονται πολύ καλύτερα Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το θέμα και συμφωνώ και με τη συνάδελφό μου ε, Ντραμπάγιοβα ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, να είμαστε ξεκάθαροι και οτιδήποτε και να αποφασίσουμε αυτή τη στιγμή για την απόσπαση των εργαζομένων, αυτό να μην καταλήξει τελικά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από κάποια χρόνια. Γιατί οι εταιρείε αλλά και οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν επακριβώ πού βρίσκονται. Η κυρία Σόιντερα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, οι αγαπητές συνάδελφοι Μωρέν Σαρτιέ και Αγκάρες είχαν πολύ δύσκολο, ε, πολύ δύσκολο έργο ε, και μάλιστα έπρεπε να παρουσιαστεί αυτό πριν από την εφαρμοστική λειτουργία, ε, οδηγία. Με συγχωρείτε. Εκτιμώ την προσπάθειά σας όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων. Ε, συμφωνώ απολύτως ότι αυτό πρέπει να γίνει. Όμως έχουμε την ευθύνη να προετοιμάσουμε την, ε, μια έκθεση που να είναι ε, αποδεκτή. και να μπορούμε να την υποβάλουμε και στα ε, κοινοβούλια των 11 κρατών μελών. Γι' αυτό θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για τις τροπολογίες που θα καταθέσω. Καταρχά θα πρέπει να εξαιρεθεί ο τομέα των μεταφορών από αυτή την οδηγία γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο και χρειάζεται μια ειδική τομεακή οδηγία, ε, η νομοθεσία. Η Κομισιόν αλλά και οι συνάδελφοι υπογράμμισαν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του τομέα των μεταφορών. Συμφωνώ με την συνάδελφο Αγνιέσκα Κοσλεβίσκα ότι αυτό ότι αυτό θέτει πολλά προβλήματα. Θα ήθελα να προτείνω λοιπόν ένα διπλό σύστημα για τους αποσπασμένους κάτω των 6 μηνών θα πρέπει να εφαρμόζεται το ισχύον σύστημα. Για τις αποσπάσεις πάνω των 6 μηνών το νέο κανόνα αμοιβών που προτείνει η Κομισιόν και οι εισηγήτριες. Αυτό το σύστημα θα είναι πιο ευνοϊκό για τις μικρές ε, επιχειρήσεις που δεν θα επιβερεθούν με υπερβολική γραφειοκρατία και φραγμούς. Ελπίζω λοιπόν ότι θα καρποφορήσει η συζήτησή μας και ότι θα βρούμε μια καλή λύση. Σας ευχαριστώ. Thank you, Κυρία Στάνρουκ, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια η οποία σε μία από τις τελευταίες συνεδριάσεις όταν αρχίσαμε να συζητάμε το θέμα ε, μας ε, παρουσίασε διεξοδικά την έκθεσή της. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που αυτή τη συζήτηση που είχε ξεκινήσει τότε την συνεχίζουμε σήμερα. Και ξέρετε να συζητάμε ψύχρεμα και νυφάλια γιατί ο στόχος τελικά αυτής της οδηγίας είναι να καλύψουμε τα κενά. Υπάρχουν παραθυράκια τα οποία ήδη από το 1996 είχαν ενταχθεί στα νομοθετήματα. Αυτά τα παραθυράκια να τα κλείσουμε, να τα εξαλείψουμε και τελικά και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τότε ε, έλαβε υπόψη του τις ενστάσεις του Κοινοβουλίου και αποφάνθηκε ε, αναλόγως. Εγώ ευχαριστώ την εισηγήτρια για την πολύ καλή έκθεση. Θα πρέπει η απόσπαση να είναι δίκαιη για όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους και για τους εργαζόμενους και για τις επιχειρήσεις και δυστυχώς ισχύει το εξή. Οι εργαζόμενοι είναι εκείνοι οι οποίοι τελικά υποφέρουν από όλους τους άλλους που προσπαθούν να παρακάμψουν τους νόμους. Θεωρώ εξάλλου ότι θα πρέπει να σεβόμαστε και τις εθνικές συλλογικές ε, συμβάσεις, δηλαδή να λαμβάνονται υπόψη όλες οι συλλογικέ συμβάσεις. Όσον αφορά τις μεταφορές, και εγώ πιστεύω ότι για τους εργαζόμενους που μετακινούνται πράγματι εκεί χρειαζόμαστε διαφορετικούς κανόνες. Όμως δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε τις ε, μεταφορές πριν επιτέλους η Κομισιόν καταθέσει μία νέα οδηγία. Οι σοσιαλδημοκράτες λοιπόν ε, θα καταθέσουν ε, τροπολογίες. Εμείς το έχουμε συζητήσει σε πάρα πολλά κράτη-μέλη και θα προσπαθήσουμε να είμαστε δίκαιοι και να λάβουμε υπόψη μας όλα τα συμφέροντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Γιαζοβιέτσκα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστώ τις ε, συνεισηγητρίες για την εκπόνηση της έκθεσης, γιατί η εκπόνηση κοινή έκθεσης για τόσο επίμαχο ζήτημα, όπως είναι η απόσπαση εργαζομένων, είναι πολύ δύσκολο θέμα. Έχω λίγο χρόνο, γι' αυτό θα έρθω στο κυρίως θέμα. Η η τροπολογία 4 βαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Ε, μετά από 24 μήνες ε, προτείνει η, προτείνει οι ε, να, να αναφερθούν οι συγκεκριμένες συνθήκες πρόσληψης. Ποιες όμως ακριβώς συνθήκες πρόσληψης, ποιες χώρες μέλους. Γιατί όταν ξεπερνούμε τις 24 μήνες απόσπασης, ε, παρόλα αυτά εξακολουθούν να εμπίπτουν στο δίκαιο της χώρας αποστολής. Δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν εδώ κενά στο δίκαιο και να μείνουν μετά το 24μηνο ε, μετέωροι και απροστάτευτοι οι εργαζόμενοι. Επίσης, ε, για ένα σύντομο χρονικό διάστημα σε ποιο δίκαιο θα εμπίπτει ε, ο εργαζόμενος σε περίπτωση που είναι σύντομη η απόσπασή του. Για παράδειγμα, ε, στην ε, Γαλλία έχουμε διαφορετική κατάσταση και έχουμε ε, πολύ ογκώδη νομοθεσία, 60 σελίδες. Πώς είναι δυνατόν οι επιχειρηματίες να γνωρίζουν το εθνικό δίκαιο κάθε φορά. Επίσης, σε ποιον θα εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία. Θα πρέπει να το ξέρουμε. Και από πότε θα αρχίζει να ισχύει το 24 μήνο. Υπάρχουν πολλές ασάφειες λοιπόν. Ε, νομίζω ότι ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιλύσει αυτές τις αμφισημίε. Επίσης, το ίδιο ισχύει με την τροπολογία 16 για τι ε, αποδοχές. Ποια θα είναι τα βασικά στοιχεία για τις αποδοχές και εκεί ε, θα πρέπει να έχουμε ουσιαστικές νομοθετικές ρυθμίσεις που δεν θα επιδέχονται παρερμηνίες. Επίσης να μην παραβιάσουμε και την αρχή της επικουρικότητας και για τις μεταφορές δεν Νομίζω δεν έχει νόημα να βιάζομαι έτσι, γιατί δεν προλαβαίνω τους ή άλλως. Ο κύριος Σούλτς για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μας προσφέρει τη δυνατότητα να έχουμε ανταλλαγή απόψεων όπου μπορούν όλοι να εκφράσουν τη δική τους την άποψη. Όσον αφορά την οδηγία περί, ε, περί απόσπασης εργαζομένων, νομίζω είναι αυτονόητο ότι πρέπει να διευκρινίσουμε λιγάκι την κατάσταση. Το θέμα είναι ότι στην εφαρμοστική οδηγία το είδαμε εκεί, ότι καλές οι προθέσεις, αλλά αν δεν ε, τις λαμβάνουν υπόψη και δεν τις εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη, ε, δεν προκύπτει τελικά σχεδόν τίποτα. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα. Και εάν ε, καταστήσουμε την απόσπαση πολύ περίπλοκη, τότε καταλαβαίνετε ότι θα βλάψουμε την ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων και ενδεχομένως και να προκύψει και μαύρη εργασία. Μεγάλο πρόβλημα αυτό. Δύο-τρία θέματα που είναι σημαντικά για μένα. Το ένα είναι το θέμα της ε, αποζημίωση των εργαζομένων. Πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους έτσι ώστε η αποζημίωση να μπορεί να οριστεί, δηλαδή λύσεις που να είναι κατανοητές και για τους εργαζόμενους και για τους εργοδότες. Κατά τη δική την άποψη, μόνο εφόσον καταλήξουμε σε έναν κατανοητό ορισμό και δεν έχουμε μια αερολογία από ορισμούς, μόνο τότε θα μπορέσουμε ε, να έχουμε ε, επί της ουσίας βελτίωση και να έχουμε και λιγότερες ενστάσεις. Το θέμα που φύγει αυτή τη ιστοσελίδα για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό δεν λειτουργεί, το είδαμε. Και γι' αυτό το λόγο ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε λιγάκι το θέμα της ε, ενημέρωσης. Και κάτι άλλο, δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά όσον αφορά τη διάρκεια της απόσπασης, είναι σημαντικό να πούμε ότι το δίκαιο της φιλοξενούσας χώρας δεν πρέπει να ισχύει ε, πολύ γρήγορα, ίσως μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Και αν όμως πάλι δεν υπάρχει σωστή ρύθμιση, μπορεί να υπάρξει και εκμετάλλευση, ανεξάρτητα αν η απόσπαση θα είναι για τη διάρκεια των 18 ή των 24 μηνών. Επειδή δεν έχω χρόνο, αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Euh, Ευχαριστώ. Επειδή είμαστε μέσα στη συζήτηση θα πω δύο-τρεις βασικές ιδέες. Η θέση του Ισάλντε, την οποία στηρίζει και, και ανέφερε και η κυρία Χλαβάγιουβα που είναι η Σκιώδης, υπάρχουν τα εξής. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και ένα μικρό το 0,4% αλλά όποιο και θα είναι η λύση, το λέω και στην Κομισιόν και σε όποιον άλλο θέλει να τα ακούσει. Αυτό θα πρέπει να είναι η λύση αυτή, να, χωρίς να δυσκολέψει και χωρίς να επιδεινώσει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Όποια λύση και αν βρεθεί. Έτσι όπως έχει τώρα στο κείμενο δεν ισχύει αυτό. Γιατί βλέπω την κυρία Μογάνη Σαχτιά ότι είμαι σκληρό να κάνει νόημα. Αλλά πρέπει να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν είμαι βέβαιος ότι δεν πήραμε το θέμα αυτό ανάποδα. Και ίσως ε, γι' αυτό θέλω να προσπαθήσω να είμαι ε, ε, συμπληρωματικός. Μιλάμε για κόστη, όμως πάντοτε θα υπάρχει ανταγωνισμός με βάση το κόστος και το κόστος της εργασίας. Αν δεν ίσχυε κάτι τέτοιο στο παρελθόν, οι Ισπανοί θα ήταν ακόμα σε σε φάση που σκαρφάλωνα στα δέντρα, ε, αλλά έχουμε μετατραπεί σε μια βιομηχανική πλούσια χώρα χάρη στον ανταγωνισμό. Και έπειτα ο κύριος ε, ε, Αρντή είπε πριν από λίγο κάτι ξεκάθαρο. Έχουν το δικαίωμα να πάνε και να μείνουν μέσα σε κοντέινερ. Αυτό είναι παράδεκτο, αλλά αυτό είναι κατάχρηση της νομοθεσίας. Γιατί να μην κλείσουμε τις ε, εταιρείε που είναι απλά μια πρόσωψη, ε, τις ψευτοεταιρείες. Γιατί να μην αυξήσουμε τους ελέγχους, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για ευρωπαϊκό έλεγχο μέσω των επιθεωρήσεων εργασίας ας πούμε. Δεν είναι βλάπτοντας την ανταγωνιστικότητα και τις ελευθερίες που θα ρυθμίσουμε το θέμα των καταχρήσεων. Ευχαριστώ πολύ, ο κ. Κάντελε. Ευχαριστώ. Έχω τρία σχόλια. Καταρχήν να σας εκφράσω κάποιες ανησυχίες και την ικανοποίησή μου. Ε, καταρχήν μιλούμε για τον προσωρινό χαρακτήρα που θα πρέπει να ρυθμιστεί. Και ε, ως προς αυτό όμως υπάρχει ασάφεια. Τι είστε ακριβώς προσωρινός χαρακτήρας. Επίσης, ε, χαίρομαι για την αντικατάσταση του κατώτατου μισθού ε, από μια άλλη έννοια. Νομίζω ότι είναι πιο δίκαιο. Επίσης, ε, η απόσπαση για μερικούς θεωρείται κοινωνικό ντάμπινγκ. Νομίζω όμως είναι μια απόλυτα νόμιμη επιλογή. Συμφωνώ όμως θα πρέπει να δούμε πώς θα την περιορίσουμε ή πώς θα την οριοθετήσουμε. Αλλά θεωρώ ότι αν περιορίσουμε υπερβολικά την απόσπαση με υπερβολικές κανονιστικές ρυθμίσεις, θα εξωθήσουμε τις ε, εταιρείε να καταφύγουν σε παράνομες ε, λύσεις. Όπως ισχύει στην περίπτωση των ψεύδο αυτοαπασχολουμένων. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι η απόσπαση και η ψεύτο αυτοαπασχολούμενοι είναι τα δοχεία. Θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε νομικά το ζήτημα, να δούμε ποιε είναι οι σωστέ νομικέ βάσεις και να εξασφαλίσουμε και σαφέστερο έλεγχο πιο ενισχυμένο για να αποφύγουμε τις ατασταλίες και να περιορίσουμε τις αμφισημίες και τις φαίες ζώνες και να συντονίσουμε και το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης. Thank you, Madam Ευχαριστούμε κυρία Λίνκεβισούτε. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Όσο βρίσκομαι στην Επιτροπή αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι προτάσεις σε σχέση με αυτή την πρόταση ήταν ανέκαθεν οι πιο δύσκολες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συζητητές γιατί έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά Κυρίως διότι οι προτάσεις αυτές ε, είναι πολύ λεπτές, πολύ ευαίσθητες για τις χώρες της Κεντρικής και της ε, Ανατολικής Ευρώπης. Πολλές από αυτές τις χώρες ε, συμπεριλαμβανομένη και της Λιθουανίας επιθυμούν να έχουν δίκαιους μισθούς Πράγμα όμω που δεν γίνεται με την απόσπαση των εργαζομένων, όταν αποσπώνται οι εργαζόμενοι οι Λιθουανοί. Αντί να τους καταβάλουν μισθούς, τους καταβάλουν κάποιες, κάποια τέλη, κάποιες εισφορέ, αλλά όχι κοινωνικές εισφορές και όχι ασφαλιστική κάλυψη. Δεν μπορεί να υπάρχει ισορροπία ε, ανάμεσα στα νέα και τα κράτη-μέλη. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ρυθμίσει το θέμα που αφορά στις συνθήκες εργασίας όσων ασχολούνται με τις εμπορευματικές μεταφορές. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό, ένα χάσμα όσον αφορά τους μισθούς τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να εργαστούμε πολύ περισσότερο για να προχωρήσει λιγάκι αυτή η οδηγία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριος Λεϊαρικ, ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ τις συνεισηγήτριες για το έργο τους. Νομίζω ότι καλούμαστε να αποφανθούμε για ένα ζήτημα γενικού συμφέροντος. Θα πρέπει ταυτόχρονα να συνδυάσουμε την ε, ελευθερία της διακίνησης ε, με την προστασία και την νομιμότητα. Δεν μπορούμε ε, στον ίδιο τόπο να έχουμε εργαζομένους από διάφορες χώρες που δεν έχουν τις ίδιες αμοιβέ, δεν διχάνουν τις ίδιες κοινωνικές προστασίες, δεν καλύπτονται από τις ίδιες συλλογικέ διαπραγματεύσεις. Και υπάρχει και αυτό το θέμα που ακροθυγώς μόνο ε, θίξαμε, το θέμα της ε, στέγασης και των συνθηκών στέγασης αυτών των εργαζομένων πολλές φορές είναι απαράδεκτες. Επίσης, δεν έχουμε μόνο τον προσωρινό χαρακτήρα και σίγουρα εδώ θα χρειαζόμασταν κάποια ελαστικότητα, αλλά μόνο προσωρινό χαρακτήρα μπορούν να έχουν οι και να αποφύγουμε κάποιον που θα είναι επανειλημμένος προσωρινός. Μπορεί να, να έρθει προσωρινά για ένα διάστημα, να επιστρέψει και να ξαναγυρίσει. Θα πρέπει να το αποφύγουμε. Και δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να αποκλείσουμε τις μεταφορές από το πεδίο εφαρμογής οδηγίας για πολλούς και διάφορους λόγους. Καταρχήν, είναι πολλά τα διακυβεύματα στις μεταφορές. Οδική ασφάλεια, περιβάλλον. Είναι πολλές οι προκλήσεις ε, από τις μεταφορές. Επίσης ε, η ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών, αλλά υπάρχουν και άλλα διακυβευόμενα. Υπάρχουν, ε, για παράδειγμα, μεγάλες επιχειρήσεις της Δυτικής Ευρώπης που χρησιμοποιούν κάποιες θηγατρικές ή εικονικές εταιρείες, εταιρείες γραμματοκιβώτιες χώρες Ανατολικής Ευρώπης ψάχνοντας οδηγούς ε, για τις μεταφορές και δημιουργώντας μία παρανομία. Θα πρέπει αυτό το τομέα να τον καλύψουμε, δεν μπορούμε να τον αφήσουμε αριθμίστο και ξέφραγο αμπέλι. Θα ήταν ε, λάθος. Επίσης, θεωρώ ότι θα πρέπει να βρούμε ένα σωστό σύστημα ελέγχου. Διερωτώ λοιπόν πως θα πρέπει να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι και να, στη, να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό σώμα επιθεωρητών εργασίας. Ευχαριστώ. Τελειώσατε, μάλιστα. Ο κύριος Ρόχβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τι ε, δύο συνεισηγητρίε και το επιτελείο των σχεδόν εισηγητών για το αξιόλογο έργο του. Θα είμαι με τριόφρον, γιατί είμαι ε, καινούριο μέλο τη Επιτροπής, οπότε μόλι ε, τώρα τελευταία να παρακολουθώ αυτό το ζήτημα, θα σα παρουσιάσω σύντομα. Καταρχήν δεν θεωρώ ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ του του νέου κειμένου ε, και της ανάγκης να εφαρμοστούν ε, τα υφιστάμενα κείμενα. Δεν νομίζω ότι είναι αντιφατικό αυτό. Είναι αλήθεια ότι το θέμα επήγει, γιατί είναι ε, μέλημά μας ε, να δημιουργήσουμε μια ασφάλεια δικαίου, γιατί το ζήτημα αυτό έχει αναστατώσει και έχει ανησυχήσει πολλούς συμπολίτες μας. Επίσης, η πατρίδα μου, η Γαλλία, θεωρείται πολλέ φορέ ω ε, χώρα που επικρίνει την οδηγία. Λάθο. Έχουμε πολλού αποσπασμένου εργαζομένου, αλλά είμαστε μια χώρα που έχει πολλούς ε, και που δέχεται πολλούς αποσπασμένους και στέλνει πολλούς αποσπασμένους εργαζόμενους. Είναι λάθος ή υπεραπλουστευμένο να θεωρείται ότι η Γαλλία είναι ενάντια της οδηγίας αυτής. Επίσης, ε, είμαστε όλοι υπέρ της ενιαίας αγοράς και της ελευθερίας διακίνησης. Ε, μόλις ψηφίσαμε για την ΣΕΤΑ, την συμφωνία με τον Καναδά. Οπότε δεν θα πρέπει ενώ δίνουμε ένα μήνυμα ανοιχτό προς τον έξω κόσμο να είμαστε ε, υπερβολικά κλειστοί και περιοριστικοί στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που με εντυπωσιάζει στο κείμενο είναι ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε το κλειδί της όλης υπόθεση που είναι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Δεν θα πρέπει να επιρρύπτουμε ή να αλληλοκατηγορούνται τα κράτη-μέλη μεταξύ τους. Θα πρέπει να δώσουμε έφαση στη συνεργασία των κρατών μελών. Αλλιώ θα υπάρχουν αντιφάσει στις δράσει του ε, και θα δημιουργηθεί ένα επικίνδυνο τοπίο. Επίση, ε, να διευκρινίσουμε το θέμα των αποδοχών που αυτή τη στιγμή είναι ασαφές. Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς μεταφορές, σας ομολογώ ότι εγώ δεν έχω αποκρισταλώσει ακόμη άποψη για το θέμα αυτό. Αν θα πρέπει η οδηγία να καλύπτει και τις διεθνείς μεταφορές. Πάντως, αν γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο σαφείς στη διατύπωση από ό,τι μέχρι στιγμής. Εγώ θα ήθελα αναφερθώ στην πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημιουργεί ένα σιδερό παραπέτασμα προκειμένου να εμποδίσει την απόσπαση εργαζομένων από τις ανατολικές χώρες στις υπόλοιπες χώρες. Νομίζω ότι θα πρέπει στόχος της οδηγίας ε, είναι να ε, μην δημιουργηθούν φαιές ζώνες και νομίζω ότι τελικά η μεγάλη χαμένη αυτής της υπόθεσης θα είναι οι νομοταγείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις που με πολύ δυσκολία τα βγάζουν πέρα είναι δύσκολο να ανταγωνιστούν τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην ε, ενιαία αγορά και θα αναγκαστούν σε κλείσιμο. Έχουμε μία οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι επιβλαβής για την ε, ενιαία αγορά και μάλιστα δημιουργεί δικαιολόγητη ε, δικαιολόγητο περιορισμό στην παροχή των υπηρεσιών, παραβιάζει ε, την ε, αρχή της επικουρικότητας, γι' αυτό και διαμαρτυρήθηκα τα κράτη-μέλη και νομίζω ότι η έκθεση δεν διορθώνει όλα, όλες αυτές τις αδυναμίες της αρχικής οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι μόνο δεν τις διορθώνει, αλλά τις οξύνει και όλα. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Χότς για ένα λεπτό γιατί ήδη μιλήσατε. Ευχαριστώ. Η οδηγία για την ε, ίση αποδοχή, για την ίση παροχή εργασίας ε, φαίνεται καλή στα χαρτιά και ίσως είναι ελκυστική ρυθμίση για το μέλλον, αλλά στην παρούσα κατάσταση ουσιαστικά δημιουργεί ε, τείχος μεταξύ Ανατολικής και, δι, και ε, Δυτικής Ευρώπης. Και νομίζω ότι έτσι θα ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας και θα οδηγήσουμε πολλές ε, πολωνικές εταιρείες στην απομόνωση, γιατί δεν θα έχουν πρόσβαση στη δυτική αγορά. Επίσης, δεν θα ευνοήσουμε την απόσπαση εργαζομένων και ταυτόχρονα παραβιάζουμε την αρχή της επικουρικότητας. Θα έχουμε τη διαδικασία της κίτρινης κάρτας. Παρόλο που πολλές χώρες ήδη έχουν εκφράσει την, τις αντιδράσεις τους και την αντίθεσή τους με την οδηγία. Το πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η αδήλωτη εργασία. Και αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε περισσότερο. Η οδηγία είναι ουσιαστικός προστατευτισμός γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση προβάλλεται α, ως απόδειξη της θεωρίας του Ντάρβιν ότι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό και ισχύει το δίκαιο της ζούγκλας. Ο ισχυρότερος κερδίζει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, καθυστέρησα γιατί ήμουνα στην αντιπροσωπεία του Μεξικού τη Δευτέρα. Πάμε στο Μεξικό και φαντάζομαι όλοι καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι αυτή η αποστολή γιατί προφανώς και οι Μεξικανοί βρίσκονται σε δύσκολη θέση και θέλουμε εμείς να τους εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας. Εγώ τώρα θα αναφερθώ σε δύο θέματα. Το, ε, το πρώτο είναι στην Most Favorite Principle, μου είπαν ότι αυτό αποτελεί ε, παραβίαση του κανονισμού Ρώμη 1. Ε, εγώ στα έγγραφά μου δεν το βρήκα. Αγαπητή Ελίζαπετ και αγαπητή Άγνες, μπορώ να φανταστώ ότι η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής το να υπάρξει μια προσθήκη, γιατί αυτό θα βοηθούσε. Κοιτάξτε, αν δεν υπάρχει άλλη νομική μορφή από του ενδιαφερόμενου. Ίσως αυτό είναι μια λύση που μπορείτε να συμφωνήσετε. Επίση, δεν θέλουμε αντιπαράθεση ανατολή δύση. Υπήρχε κάποτε, αλλά δεν θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η αντιπαράθεση και γι' αυτό πράγματι θέλουμε να ε, καταπολεμήσουμε την αδήλωτη εργασία. Στη δική μου τη χώρα τη Γερμανία είμαστε πολύ πιο σκληροί από άλλε χώρε. Ακριβώ για να ε, διασφαλίσουμε την δικαιοσύνη στι ε, θέσει απασχόληση και στην εργασία. Το άλλο, την ιστοσελίδα ε, που το απαντήσατε την προηγούμενη φορά πολύ σωστά κατά την άποψή μου στις τροπολογίες 14 και 21 υπάρχει το θέμα των αντιπροσωπευτικών συλλογικών ε, συμβάσεων δηλαδή μια πρόταση να επεκτατεί η ισχύς και σε αντιπροσωπευτικές συλλογικέ συμβάσει. Οι νομοματείς μου είπαν ότι είναι μια, ένας νέος όρος που δεν έχει διευκρινιστεί ε, σε νομικό επίπεδο. Η δική σας άποψη ποια είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ότι είσαστε ανοιχτοί και διαφανείς. Είχαμε πάρα πολλούς ε, καλούς ε, διμερείς διαλόγους. Επιτέλους, το βρίσκω πολύ σημαντικό αυτό. Ο κύριος Μπροκ για δύο λεπτά. Και εγώ ευχαριστώ. Λίγες παρατηρήσεις θα κάνω και θέλω και εγώ να ευχαριστήσω ε, τις εισηγήτριες. Κάποιοι, κυρίως από την Ανατολική και την Κεντρική Ευρώπη, κάνουν λόγο για απομόνωση. Νομίζω πρέπει να είναι σαφές ότι η Ευρώπη δεν είναι εργαλείο για να μπορέσει να παρακάμψει κανείς κοινωνικές διατάξεις και εργασιακές ρυθμίσεις. Κάθε άλλο. Ε, δεν είναι δυνατόν λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάποιες χώρες οι ε, συνθήκες εργασίας να επιδεινώνονται, γιατί αν ισχύει αυτό, τότε τα πράγματα σημαίνει ότι φτάσαμε στο τέλος. Άρα δηλαδή αυτό που μας ενδιαφέρει είναι προστασία των εργαζομένων σε φιλοξενούσες χώρες αλλά και προστασία των εργαζομένων από τις χώρες προέλευσης. Και αυτός ο κανονισμός δεν προστατεύει τους εργαζόμενους από τις χώρες προέλευσης. Και να σας πω το εξή. αν το τι γίνεται στη δική μου την πατρίδα διαπιστώνω ότι πολλοί οδηγοί φορτηγών το Σαββατοκύριακο το περνάνε στη Γερμανία σε πάρκινγκ και χώρους στάθμευσης στη Γερμανία. Ζουν εκεί ε, με απαράδεκτες συνθήκες και οι άνθρωποι αυτοί ε, έχουν ε, αποδοχές που είναι επίσης απαράδεκτες. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν επιδείνωση και των ιδίων των ανθρώπων και όλων των άλλων που εργάζονται όμως στη Γερμανία. Ως εκ τούτου, αυτές οι προϋποθέσεις που δέχονται οι φιλοξενούμενοι εργαζόμενοι, αυτές οι προϋποθέσεις και αυτοί οι όροι δεν είναι σωστοί. Δεν είναι οι όροι ε, που θα πρέπει να επιτρέπονται σε μια κοινωνική Ευρώπη. Γιατί η ανταγωνιστικότητα μπορεί να διασφαλιστεί και με άλλους τρόπους και όχι με αυτούς, τους απαράδεκτους. Η κυρία Ντέλη. Είναι εδώ. Η κυρία Λαουριστίν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω δεν είναι σωστό να μιλάμε εδώ για Ανατολή και Δύση, γιατί και στην Ανατολή δεν είναι όλοι οι ίδιοι και εκεί υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση. Εγώ, ας πούμε, έρχομαι από την Εστονία. Το βασικό μας πρόβλημα είναι η σχέση με τη Φινλανδία. Εστονία, Φινλανδία, αυτό είναι το πρόβλημα. Ε, βέβαια έχουμε πολύ καλή συνεργασία και δεν έχουμε τα προβλήματα που τίγεται. Αλλά θέλω να επισημάνω κάτι άλλο, ότι με αυτές τις συλλογικέ συμβάσεις, τις ευρύτατες, δημιουργείται μια λυσίδα με λιγότερη διαφάνεια από συμφωνίες ε, που είναι μεγαλύτερης εμβέλειας. Γι' αυτό λοιπόν για τους δικούς μας τους εργαζόμενους και τους πολίτες είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσουν ε, όλες αυτές τις πληροφορίες. Ως εκ τούτου ζητάνε από τις εταιρείε ε, να βελτιώσουν τις συνθήκες. Όσοι έχουν τώρα τα πράγματα εμείς λέμε ότι υπάρχει αδικία. Αυτές οι μεγάλες εταιρείε δεν είναι ανοιχτέ και για τους εστονούς, για τους δικούς μας ανθρώπους είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκτήσουν ε, όλες αυτές τις ε, πληροφορίες. Ο κ. Φουντούλης, παρακαλώ. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η απόσπαση σαν ειδική μορφή απασχόλησης στηρίζεται αρχικά στην ελεύθερη παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών. Είναι ένα εργαλείο το οποίο όμως χρησιμοποιούν κατά κόρον μεγάλες εταιρείες. Ε, σύμφωνα με την Επιτροπή, ο τομέας των κατασκευών αντιπροσωπεύει το 43,7% ενώ η απόσπαση στον τομέα της μεταποίησης, της εκπαίδευσης και της υγείας είναι σημαντικές. Το θέμα των αμοιβών για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι πρέπει να αμείβονται όπως και οι εργαζόμενοι στις χώρες που απασχολούνται. Για ίση εργασία να ισχύουν ίσες αμοιβές. Ένας εργαζόμενος παραδείγματος χάρη στις κατασκευές για το ίδιο έργο λαμβάνει ίση αμοιβή με τον εργαζόμενο στη χώρα που βρίσκεται ή γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από μεγάλες εταιρείες που θέλουν μειώνοντας το μισθολογικό κόστος να έχουν περισσότερα κέρδη. Ένας επιστήμον ιατρός που ασχολείται με την έρευνα, αποσπασμένος σε μια άλλη χώρα, θα αμείβεται το ίδιο ή οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες θα μειώνουν το εργασιακό κόστος αυξάνοντας τα κέρδη τους. Στις χώρες όπως η Ελλάδα που είναι σε μνημόνιο και οι συλλογικές συμβάσεις έχουν απαξιωθεί, ποιος θα προστατεύσει τους εργαζόμενους που αναζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και αποσπώνται σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Η οδηγία θα δεσμεύσει τις επιχειρήσεις στα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ. Thank you. Mr. Christensen. Σας ευχαριστώ, κύριος Κρίστενσεν. Φου Φόρμαν, det her er jo et meget sensitivt øh, område, og det må Έχω, ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω μια λεπτή ερώτηση. Είναι πολύ λεπτό το ζήτημα και δεν θα πρέπει όντως να οδηγήσει σε ένα ρήγμα Ανατολής με Δύση. Πιστεύω ωστόσο πως οι συγγήτρες έχουν βρει καλή ισορροπία σε αυτή την έκθεση και ξέρω πως είναι πολύ δύσκολη η εξέβρεση ισορροπίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε αποσπασμένους εργαζόμενους. Όχι. Πρόκειται για ανθρώπους που έρχονται. Ο Τόμας Μαν και ο Έλμαρ Μπρόκ το είπαν ότι πρέπει να προστατευτούν αυτοί οι εργαζόμενοι ώστε να χαίρουν τον ίδιο συνθηκών με τους εργαζόμενους της χώρας υποδοχής. δεν χαίρουν λοιπόν τις ίδιες ε, κάλυψεις με τους υπολείπους που πληρώνουν τους φόρους και χαίρουν και τις κοινωνικές τους ασφάλισεις Να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για όλους, διεθνείς και μη διεθνείς εργαζόμενους. Γιατί το δύσκολο είναι να δούμε τι συμβαίνει με αυτόν τον κόσμο που πηγαίνει να έρχεται. Γι' αυτό και είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός πλαισίου συνθηκών, ορίων, κανόνων που εξασφαλίζουν ακριβώς ότι οι εργαζόμενοι, οι μετακινούμενοι χαίρουν των ίδιων ακριβώς συνθηκών. Δεν θέλουμε κανείς να μείνει εκτός κάποιες συγκεκριμένες περιοχές και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Χρειάζεται μεγαλύτερος ανταγωνισμός ανάμεσα στις εταιρείε, αλλά δίκαιος, θεμητός ανταγωνισμός και ανάμεσα στους εργαζόμενους. Ευχαριστώ. Thank ε, ευχαριστώ. Η Κάρη Μαντέλη δεν έχει έρθει. Η κυρία Γλαβάγεβα ζήτησε και πάλι το λόγο. Ναι, θα είμαι σύντομη, θα μιλήσω τσεχικά. Ε, Ζητώ συγγνώμη που ζήτησα που έκανα έκκληση. Δεν είναι μαύρο-άσπρο το θέμα εδώ. Μιλάμε για συνθήκες εργαζομένων, για στέγαση, για καταχρήσεις και τονίζουμε μόνο τα αρνητικά στοιχεία. Αλλά η απόσπαση των εργαζομένων η ίδια, αυτή καθ' αυτή, δεν είναι αρνητική, είναι θετική, όπως είναι και η ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων και υπηρεσιών. Πάντοτε υπάρχουν άνθρωποι που δεν σέβονται τους κανόνες και βρίσκουν τρόπους να τους παρακάμπτουν ε, αν αυτό θέλουμε να το καλύψουμε μέσω διοικητικών ποινών θα τιμωρήσουμε τελικά μόνο αυτούς οι οποίοι τηρούν τους κανόνες. Θέλουμε εμείς να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτούς που δεν τηρούν τους κανόνες. Δεν θα α, α, καλυτερέψει η κατάσταση μόνο επειδή θα έχουμε αυστηρότερους κανόνες. Ας μιλήσουμε απλά και μόνο για το τι είναι θετικό και τι είναι αρνητικό. Κάνω έκκληση σε όλους και πάλι. Φαίνεται σαν να μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι μόνο η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην Δύση και στην Ανατολή. Είναι, δείχνει και τη διαφορά ανάμεσα σε όσους έχουν εργαστεί σε ιδιωτικές εταιρείες και σε όσους δεν έχουν εργαστεί σε ιδιωτικές εταιρείε. Ναι, να πω και εγώ ίδια δύο λόγια. Ε, ε, να ευχαριστήσω τις εισηγήτριες, κυρία Γιουγκάριους και κυρία Μωρέν Σαρτιέ. Κάνατε εξαιρετική δουλειά μέχρι τώρα. Είναι υποχρέωση να αναζητήσουμε κάτι ε, συγκεκριμένο κάτι που να μπορεί να περάσει από το σύστημα και να δώσει και καλά αποτελέσματα. Επίσης με χαρά βλέπω την πρόταση για επέκταση της νομικής βάσης. Αυτό είναι θετικό, ένα σημαντικό βήμα για να εξασφαλίσουμε ότι η μετακίνηση, η επόσπαση μάλλον των εργαζομένων αντιμετωπίζεται στο νομικό σύστημα όπως αρχικά αυτό είχε ε, επινοηθεί με τον αρχικό στόχο δηλαδή, δηλαδή ανάπτυξη εσωτερική αγοράς. Αυτό το στόχο είχε η νομοθεσία η αρχική και η ευρύτερη νομική βάση, εάν υπήρχε από την αρχή, δεν θα έχουμε τώρα τα ίδια προβλήματα όπως τώρα, όπως τις υποθέσεις ε, Λαβάλ και τα λοιπά. Ε, δίκαιος ή αμοιβή επίσης είναι εξαιρετική σημαντική νομοθεσία μαζί με την νομική βάση, γιατί καλύπτει μια μεγάλη σειρά προβλημάτων και νομίζω πως πραγματικά ε, τα αντιμετωπίζουμε κατάματα τα προβλήματα. Απλά ήθελα να το πω γιατί είναι ένα από εκείνα που με απασχολούν στην πολιτική ε, εδώ και 10-15 χρόνια. Πιστεύω λοιπόν πραγματικά ότι κάνατε πολύ καλή δουλειά και χωρίς να διχάσουμε την Ανατολή με τη Δύση ή τους σοσιαλιστές με τους, ε, τους ε, χριστιανοδημοκράτες. Όχι. Θέλουμε να ε, κάνουμε μια καλή νομοθεσία στο να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους. θέλετε ίσως να κλείσετε και χρειάζεται χρόνο γι' αυτό. Εάν δεν χρειάζεστε όλο το χρόνο μπορούμε να δώσουμε και ένα-δύο λεπτά ίσως στην Κομισιόν και στον εκπρόσωπό τη. Ο κύριος Περέιρα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, α, ναι, παρακαλώ. Αν μπορείτε να σχολιάσετε λοιπόν το θέμα εν συντομή και μετά να το ξαναδώσουμε το λόγο στους εισηγητές. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θα περιοριστώ σε λίγα σχόλια ε, ξεκινώντας με κάποια πράγματα που μπορεί να φαίνονται αυτονόητα, αλλά καλό είναι να τα επισημαίνουμε. Καταρχήν, δεν είναι η οδηγία που δημιούργησε τις αποσπάσεις. Η απόσπαση είναι απόρρια της ελεύθερης ε, παροχής υπηρεσιών, της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών. Είχαμε απόσπαση και αποσπάσεις και πριν την οδηγία και γι' αυτό συντάξαμε την οδηγία για να ρυθμίσουμε το θέμα της απόσπασης. Οπότε η κατάργηση της οδηγίας δεν θα επηρεάσει ε, την πραγματικότητα των αποσπάσεων, γιατί η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών είναι κατοχυρωμένη στις ιδρυτικές συνθήκες. Επίσης, όπως είπαν κάποιοι ευρωβουλευτές, ε, η πιο ε, φυσιολογική και συνηθής μορφή δεν είναι η απόσπαση, αλλά η ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων. Άρθρο 45 της συνθήκης, η συμμεταχείριση με τους ντόπιου εργαζομένους και το καθεξής. Είναι μια άλλη μορφή κινητικότητας η απόσπαση, πολύ ιδιαίτερη, που εξυπηρετεί την επιχείρηση στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών. Σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας 96, ε, και εδώ θα πρέπει να είμαστε σαφείς, η οδηγία του 96 ισχύει για όλου ε, του τομεί δραστηριοτήτων. Αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα, καθαρά και εξάστερα στην, ομιλία, ε, στην οδηγία με εξαίρεση την εμπορική ναυτιλία. Και το θέμα αν οι οδικέ μεταφορέ καλύπτονται έχει ρυθμιστεί. Καλύπτονται. Φυσικά όλοι οι τομεί καλύπτονται και αναφέρεται και στην εταιρική σκέψη 10 τη ε, πρόταση. Βέβαια αναγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα των μεταφορών και η ανάγκη κάποιων προσαρμογών που θα πρέπει να γίνουν για το συγκεκριμένο τομέα, αλλά είναι σαφές ότι ο τομέας των μεταφορών καλύπτεται από την οδηγία και καλύπτεται στο μέτρο που ε, εφαρμόζει τις αποσπάσεις, όπως και άλλοι τομείς δραστηριοτήτων. Όλες ε, οι διεθνείς μεταφορές δεν συνιστούν απόσπαση και η διέλευση από την επικράτεια ενός κράτους μέλους ή η φόρτωση-εκφόρτωση δεν είναι παροχή υπηρεσίας με την έννοια ε, της απόσπασης ε, όπως την ε, ρυθμίζει η οδηγία. Και υπάρχουν στο κείμενο κάποια όρια, αλλά γενικώ το τομέας των μεταφορών καλύπτεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη είχε αναγγείλει κάποιες διευκρινήσεις που θα γίνουν ε, για τις μεταφορές ειδικά στα πλαίσια της δέσμης μέτρων για τις οδικές μεταφορές που έχουν εξαγγελθεί για τα τέλη του εξαμήνου. Επίσης, ε, υπάρχει επιτακτική ανάγκη ασφάλειας δικαίου για τον κλάδο. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις ε, ποιο είναι το ισχύο δίκαιο, θα πρέπει οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τι ρυθμίσεις ισχύουν σε περίπτωση απόσπασης. Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε αυτή την κατάσταση και το γεγονός ότι η οδηγία του 1996 δεν ήταν και πολύ αποδοτική από αυτήν την άποψη. Και η έννοια των ελάχιστων συντελεστών αποδοχών δεν είναι ε, σαφής. Το αντίθετο και απόδειξε η νομολογία του ΔΕΚ που τις περισσότερες φορές μπορεί να ευνηδίασε, αλλά αποδεικνύει ακριβώς ότι στην πράξη ήταν ασαφής ορισμός και άρα δεν ήταν εύκολη η εφαρμογή του. Στην πράξη, οι επιθεωρητές εργασίες στις περισσότερες χώρες υποδοχής ερμηνεύουν την έννοια του ελάχιστου συντελεστή μισθού ε, με την ε, έννοια του ελάχιστου μισθού, του κατώτατου μισθού. Δεν είναι το ίδιο κατώτατο συντελεστή και κατώτατο μισθό. Αλλά η έννοια αυτή είναι προσδιοριστή, δεν, προσδιορι... δεν ε, ορίζεται στα εθνικά δίκαια, γι' αυτό και δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου. Και μερικές φορές συγχαίεται με την έννοια του κατώτατου μισθού. Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε αυτή την έλλειψη ασφάλεια δικαίου που υπάρχει και την ανάγκη σαφήνεια. Βέβαια, η δική μα πρόταση είναι πιο σαφή για τι αμοιβέ. Αναφέρονται κάποια υποχρεωτικά στοιχεία για του ε, ε, εθνικού εργαζομένου. Και θα πρέπει ε, να γνωρίζει και η επιχείρηση και ο εργαζόμενος σε κάθε χώρα υποδοχής ποια είναι τα βασικά στοιχεία που αποτελούν το, την αμοιβή. Αυτό διευκολύνει και τους επιθεωρητές εργασίας. Και θα πρέπει ε, και να το λαμβάνω αυτό υπόψη και οι συλλογικέ διαπραγματεύσει. Να γνωρίζουν ποια είναι τα, πραγματικά, τα υποχρεωτικά στοιχεία και ποια όχι. Νομίζω ότι αυτή η διευκρίνηση γίνεται ακριβώ για να διευκολύνει το έργο των επιθεωρητών εργασία στη χώρα υποδοχή. Μπορεί κάποιο να διαφωνεί πολιτικά, αλλά από άποψη ασφάλεια δικαίου ήταν απαραίτητη αυτή η διευκρίνηση. Και τέλο, να και ήδη μακρηγόρησα, να αναφερθώ σε κάποιε κόκκινες γραμμές που δεν θα πρέπει να υπερβούμε. Οι κόκκινες αυτές γραμμές που είναι ανυπέρβλητες είναι το γεγονός ότι επιβάλλουμε σε επιχειρήσεις που κάνουν αποσπάσεις, ε, επιβάλλουμε διατάξεις που δεν θα ίσχυαν για τις, τοπι... για τις ε, τοπικές επιχειρήσεις, για τις ντόπιε επιχειρήσεις. Αυτό θα ήταν αντίθετο και προς την οδηγία και προς το σκοπό που επιδιώκει η οδηγία, αλλά αντίθετο και προς τις συνθήκες και οι συμφωνίε συλλογικών διαπραγματεύσεων δεν μπορεί να ε, περιλαμβάνουν κανόνε που δεν ισχύουν γενικώ ή που δεν ισχύουν για τι επιχειρήσει ε, τη περιφέρεια, ε, τη χώρα ή του κλάδου. Κάτι τέτοιο θα συνιστούσε διάκριση ει βάρο των διασυνοριακών υπηρεσιών και θα δημιουργούσε πολλές, θα δημιουργούσε πολλές αμφιβολίες ως προς την αμοιμότητα τη πρόταση. Τέλο για το θέμα των αμοιβών και την ανάγκη που επισήμαναν πολλοί για καλύτερο ορισμό αυτής της έννοιας, θα ήθελα να σας πιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι όπως και η προηγούμενη έννοια που ανέφερα στην οδηγία του 96 του ελάχιστου ποσοστού α, μισθού, ε, ο προσδιορισμός του μισθού της αμοιβή εναπόκειται στα κράτη-μέλη. Κάτι τέτοιο υπερβαίνει τι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και σε μια Ευρωπαϊκή Οδηγία περιλαμβάναμε ορισμό για ε, το τι εστί σε εθνικό επίπεδο αμοιβέ ήταν ε, παράνομο. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της χώρας υποδοχής να ορίσει τι εστί αμοιβή και δεν θα πρέπει να πέσουμε σε αυτή την παγίδα, γιατί έτσι θα παραβιάζαμε την αρχή της επικουρικότητας. Δεν λέω ότι δεν θα μπορούσαμε να επεξεργαστούμε κάπως καλύτερα το κείμενο και να διορθώσουμε ίσως τη διατύπωση, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε την αμοιβή. Κάτι τέτοιο να πόκειται στο κράτος μέλος υπόδοχης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τώρα θα πάρουν το λόγο οι εισηγήτριες. Κυρία Ιονγκέριος και μετά η κυρία Μαρέν Σαχτιά. Um, ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ επίσης και όλους τους ε, συναδέλφους για αυτή τη συζήτηση η οποία πράγματι ε, αρκετές φορές είναι φορτισμένοι συναισθηματικά και αυτό είναι λογικό γιατί η ελευθερία της μετακίνησης ε, προκαλεί πολλές συζητήσεις σε όλα τα κράτη-μέλη. Ε, πάντως νομίζω ότι αν θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδος και νομίζω αυτό το θέλουμε όλοι μας τότε πρέπει να παραγωνίσουμε τα συναισθήματά μας, να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει και να εντοπίσουμε τα κενά στο σύστημα για να δούμε τι είδους αγορά εργασίας επιθυμούμε να αποκτήσουμε. Η Ελίζαμπετ αλλά και η Νέλη ε, είπαν το ίδιο ότι παράλληλα με την ελευθερία της μετακίνησης πρέπει να την ελευθερία διακίνηση υπηρεσιών είναι πολύ σημαντική η ελευθερία μετακίνησης των εργαζομένων. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι για μένα προσωπικά η ελευθερία μετακίνηση των εργαζομένων είναι και δικαίωμα των εργαζομένων, το οποίο και θα υπερασπιστώ σε οποιαδήποτε συζήτηση και αν λάβει η χώρα. Αν λοιπόν γνωρίζουμε ότι επ' αυτού συμφωνούμε όλοι, ότι πραγματικά θέλουμε να υπερασπιστούμε αυτό το βασικό δικαίωμα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τους εργαζόμενους και για τις επιχειρήσεις, ε, τότε είναι σημαντικό για μας ε, να δούμε ποια, τι είναι η αρχική οδηγία, πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση και πώς ακριβώς ε, θα μπορέσουμε να βρούμε νέες και σύγχρονες απαντήσεις για προβλήματα που υπάρχουν στην αγορά εργασίας. Χαίρομαι πάρα πολύ που και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τοποθετήθηκε επί ορισμένων θεμάτων γιατί για μένα ξέρετε είναι σημαντικό να οριστεί το θέμα των αποδοχών. Για μας είναι σαφές. Οι αποδοχές ορίζονται από τα κράτη-μέλη. Και αυτό το έχουμε καταγράψει σε μία από τις ε, τροπολογίες μας προς μία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ίσως μπορεί να υπάρξει κάποια βελτίωση, αλλά εν πάση περιπτώσει οι αποδοχές ορίζονται από τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι σημαντικό. Και από ό,τι άκουσα θα υπάρχει και ένα σχετικό έγγραφο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν ξέρω, ίσως για το Συμβούλιο, έτσι είχα ακούσει. Και αυτό ίσως βοηθήσει εκείνους τους συναδέλφους οι οποίοι αναζητούν τον ορισμό των αποδοχών. Αλλά πρέπει να είναι σαφές όπως σας είπα, ότι οι αποδοχές ορίζονται πάνω απ' όλα από τα κράτη-μέλη. Ορισμένοι συνάδελφοι έκαναν σχόλια για το θέμα της ε, στέγασης. Και εγώ λοιπόν ε, σκέφτομαι να καταθέσω κάποιες προτάσεις από αυτού. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι για έναν αποσπασμένο εργαζόμενο αυτοί οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι δεν πρέπει να ε, καταβάλουν οι ίδιοι τις δαπάνες διανυκτέρευσης και μετακίνησης. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το εξετάσουμε στην επόμενη φάση όπου θα εξετάσουμε την έκθεση. Ε, αυτά που ελέγχθησαν για τις μεταφορές, αυτά θα είχα πει και εγώ ότι αυτή η οδηγία καλύπτει τι όλους τους τομείς εκτός από τη μετακίνηση μέσω θαλάσσης. Και εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ ε, να έχει διευκρινίσει ακριβώς η Επιτροπή τι ακριβώς περιλαμβάνει η πρότασή της ε, για τους ε, μετακινούμενους, έντονα μετακινούμενους εργαζόμενους και να ξέραμε και πώς θα αντιδράσει και το Συμβούλιο. Θα ήταν όλα πάρα πολύ ωραία. Όμως όλα αυτά δεν είναι σαφή, είναι κάτι που θα πρέπει να το εξετάσουμε στο μέλλον και τώρα θα πρέπει εδώ να είναι απόλυτα σαφές ότι αν δεν υπάρξουν ε, νέοι κανονισμοί για τους ε, συχνά μετακινούμενους εργαζόμενους θα πρέπει εμείς να τους προστατεύσουμε. Για μένα λοιπόν η συζήτηση ήταν πλούσια και προσβλέπω σε προτάσεις που θα κατατεθούν για να βελτιωθεί η έκθεση. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι καθήκον όλων μας. Δηλαδή να καταλήξουμε σε μια καλύτερη έκθεση με ευρύτατη βάση χωρίς να υπάρχουν κενά εδώ από την Επιτροπή μας που θα φανούν αργότερα στην Ολομέλεια. Μου αρέσουν οι τροπολογίε και οι συζητήσεις αρχής ε, κατά καιρού, αλλά όσον αφορά αυτό το θέμα νομίζω ότι θα πρέπει να ε, παραμείνουμε νυφάλιοι και με νυφαλιότητα να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Κυρία Μωρέν σωτιά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα πρώτα λόγια μου είναι οι ευχαριστίες μου στην Αγνές Ιουγκάριους, με την οποία συνεργάστηκα με μεγάλη, μεγάλο, μεγάλη όρεξη για αυτό το θέμα. Ναι, συζητήσαμε γιατί ανήκουμε σε δύο διαφορετικές πολιτικές ομάδες, αλλά ήδη η έκθεση αυτή είναι ένα πρώτο βήμα μπροστά στην οικοδόμηση μιας κοινή πλατφόρμας, ενός κοινού οράματος για το τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να ρυθμίσουμε το πρόβλημα των αποσπασμένων εργαζομένων. Και βεβαίως θέλω να ευχαριστήσω το σύνολο των σκιωδών εισηγητών ή να τους επιβεβαιώσω ότι βεβαίως η πόρτα μας ε, είναι πάντοτε ανοιχτή για να εμβαθύνουμε τις συζητήσεις ε, τέτα τέτ. Είμαστε αποφασισμένες να καταλήξουμε σε κείμενο. Είναι ευθύνη μας κοινή κάθε πολιτική ομάδα, μάλλον καμιά πολιτική ομάδα δεν έχει δει το δικαίωμα να αποτύχει σε αυτήν την αναθεώρηση ενός κειμένου που είναι πια 20 ετές και δεν ανταποκρίνεται στη σημερινή πραγματικότητα. Να ευχαριστήσω και το σύνολο των συναδέλφων που συμμετείχαν στη σημερινή συζήτηση, κυρία Πρόεδρε, διότι είναι σπάνιο να έχουμε τόσους συναδέλφους που να θέλουν να ε, συμβάλλουν με τη δική τους πολιτική άποψη και την εθνική τους πολιτική άποψη συχνά για το τι ε, αντιπροσωπεύει λοιπόν για τους ίδιους αυτό το θέμα. Να πούμε λοιπόν ότι αυτή η οδηγία αφορά τους αποσπασμένους εργαζόμενους και όχι τους υπόλοιπους. Οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι είναι ε, μια ειδική κατηγορία. Δεν μιλάμε ας πούμε για τους ε, γιατρούς που είναι ελεύθεροι επαγγελματίε, ελεύθερο επάγγελμα. Είναι άλλο. Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή αυτής της οδηγία. Εστιαζόμαστε λοιπόν σωστά στο θέμα μα για να επιτύχουμε την εργασία μα. Δεύτερη μου παρατήρηση θα έλεγα Προσοχή, προσοχή στις στατιστικές. Ξέρω ότι όταν μιλάμε και συσχετίζουμε τον αριθμό των αποσπασμένων εργαζόμενων στον αριθμό των συνολικών των εργαζομένων είναι ένα μικρό κομμάτι τους. Όμως έχουμε το δικαίωμα όταν μιλάμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να πούμε ότι είναι αυτοί λίγοι άστε, δεν, δεν μας απασχολούν. Όχι, δεν το έχουμε αυτό το δικαίωμα. Όμως αυτό που είναι το πραγματικό πρόβλημα και που δεν το δείχνουν οι στατιστικές ε, είναι ότι ο αριθμός των αποσπασμένων εργαζόμενων ποικίλει σε τεράστιο βαθμό ανάλογα με το τομέα δραστηριότητας. Και οι κύριοι τομείς που είναι οι οικοδομές, η γεωργία, οι επιχειρήσεις και οι μεταφορές, εκεί οι στατιστικές σας ε, δεν αξίζουν ε, διάρα. Μην πιστεύετε λοιπόν ότι οι εμπειρογνώμονες είναι πάντοτε ε, τίμοι. Εγώ ε, δούλεψα ε, πάρα πολύ για αυτά τα θέματα και μου αρέσει πολύ η ακρίβεια στην ανάλυση. Τρίτη παρατήρηση. Θελήσαμε να σεβαστούμε την επικουρικότητα των κατών μελών όσον αφορά τον καθορισμό των αποδοχών και δέχομαι και λέω αυτό που είπε η Κομισιόν και η Αγνές ότι ναι είμαστε λιγότερο συνηθισμένοι σε αυτό αλλά νομικός είναι πραγματικά πολύ συγκεκριμένο και ξεκάθαρο και έχουμε και γνωρίζουμε σε τι αντιστοιχεί αυτό. Αν λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι χρειάζεστε περισσότερες νομικές πληροφορίες για αυτό το σημείο, είμαστε απολύτως έτοιμοι να σας τις δώσουμε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πάντως δεν θα καταφέρουμε τίποτα εάν βγούμε από το ευρωπαϊκό μας πνεύμα το οποίο ε, το έχουμε κοινό για να μπούμε σε ένα έναν διχασμό Ανατολή-Δύση. Όχι. Εγώ δεν το έχω καθόλου αυτό στο μυαλό μου και καμία απολύτω θέληση δεν έχω να γίνει κάτι τέτοιο. Είμαι έντιμη και οφείλω να σας πω ότι γνωρίζω την διαφορά της κατάστασης που επικρατεί ανάμεσα στους μεταπροσπασμένους, στις επιχειρήσεις, το τι γίνεται ανάμεσα σε Ανατολή και και δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε προκαθορισμένα πλαίσια ούτε να είμαστε δογματικοί. Σας ε, θερμοπαρακαλώ, η εργασία μας θα πρέπει να εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πνεύμα. Να διαπνέεται μάλλον από ευρωπαϊκό πνεύμα. Δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα είπε η Αγνές. Θέλω απλά να προσθέσω σε αυτά. Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο, το οποίο πρέπει να το πιάσουμε από τα μαλλιά γιατί είναι αυτές οι διάφορες ε, υπεργολαβίες στην αλυσίδωτά. Δηλαδή, αποσπασμένος από την εταιρεία, στην τάδε εταιρεία, μετά στην άλλη εταιρεία, μετά ε, παρακεί, παρακεί. Ε, και αυτό θολώνει τα νερά και δεν μπορεί να υπάρξει πλέον έλεγχος, όπως θέλει η Ντανούτα να βάλει στην οδηγία την εκτελεστική. Εκεί σε αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ε, συγκεκριμένοι, να μην υπάρχει απόσπαση αλυσιδωτή μέσα σε άλλες δηλαδή εταιρείες που αναλαμβάνουν τις υπεργολαβίες. Έπειτα, Έχουμε πίσω μας ε, γενναίες ε, νέων του Έρασμος που έχουν συνηθίσει να εκπαιδεύονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ένα ευρωπαϊκό πνεύμα. Δεν πρέπει να μείνουμε στο παρελθόν. Πρέπει να προετοιμάσουμε τη μελλοντική γενιά. Και τέλος ε, να σας πω ότι πρέπει να οικοδομήσουμε και την βάση της κοινωνικής Ευρώπης ότι το ραντεβού του 2019 για τις ευρωεκλογέ θα παιχτεί στο, πάνω σε αυτό το θέμα της Ευρώπης των πολιτών και θα ήθελα όλοι μαζί να έχουμε συμβάλει με το λιθαράκι μας σε αυτή την Ευρώπη που είναι η Ευρώπη του μέλλοντος, η Ευρώπη των Ευρωπαίων ε, πολιτών. Και τέλος οι και εγώ αποφασίσαμε ένα πράγμα κυρία Πρόεδρε ότι η εκθεσή μας θα σας δώσει το νομοθετικό αποτύπωμα, δηλαδή δεν είμαστε υποχρεωμένοι, αλλά επιλέξαμε να το κάνουμε, θα έχετε τον κατάλογο όλων όσων συναντήσαμε. Ε, συνδικάτα, εργοδότες, λόμπι, κλάδι επαγγελματική, θα ξέρετε τα πάντα όσον αφορά τα παρασκήνια της εργασίας μας. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Γεσοβιέτσκα, σύντομα, παρακαλώ. Θα ήθελα, Ελίζαμπετ, ε, ελπίζω να μην μεταφράστηκες καλά, γιατί, επαναλαμβάνω, ελπίζω να μην ε, μεταφράστηκες καλά, αλλά εγώ κατάλαβα από αυτά που άκουσα, ε, ότι είπες ότι θέλεις ε, στα πλαίσια της οδηγίας ε, ε, για την εφαρμογή να περιλαμβάνεις κάποια στοιχεία για την απόσπαση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ντανούτα, δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα ότι θα θέλαμε να μην υπάρχει από αλυσιδωτή απόσπαση όταν δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το εφαρμοστέο εργασιακό δίκαιο για τους εργαζομένους. Οπότε, στο σχέδιό μας λέμε σε περίπτωση αλυσιδωτής απόσπασης, για να είναι σαφές, ισχύει το δίκαιο της χώρας υποδοχής όχι το δίκαιο της χώρας που βρίσκεται το Γραφείο Μερικής Απασχόλησης, το δίκαιο της χώρας υποδοχής. Αυτό που είπα και σε αυτό αναφέρθηκα ε, γι' αυτό είπα ότι αναφέρθηκα στην οδηγία, θέλεις να γίνουν έλεγχοι, γιατί για να τεθεί σε εφαρμογή δική οδηγία θα πρέπει εμείς εκ των προτέρων να ορίσουμε τα στοιχεία και τους όρους αυτού του ελέγχου για να μπορέσει να εφαρμοστεί μετά η οδηγία για την οποία εσύ είσαι αρμόδια. Αυτό είπα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ στην προηγούμενη συνεδρίαση όταν ζήτησα να αναβληθεί η συζήτηση για να έχουμε περισσότερο χρόνο για τη συζήτηση ε, είχαμε συμφωνήσει να έχουμε τρία λεπτά καθένα. Σήμερα το αλλάξατε. Όταν γίνονται τέτοιε αλλαγέ, θα ήθελα να μα ενημερώνει εκ των προτέρων η γραμματεία. Γιατί για πολλού από εμά το δίλεπτο είναι πολύ λίγο χρόνο. Και μα έμεινε μισή ώρα μέχρι το τέλο. Θα μπορούσαμε να είχαμε εκμεταλλευτεί και αυτό το υπόλοιπο μισάωρο και αντί για δίλεπτο να μιλούσε τρίλεπτο καθένα. Θα ήθελα να ενημερωνόμαστε και των προτέρων άλλε φορέ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι λεπτομέρειε και το πώ αποφασίστηκε αυτό. Αλλά νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι θέλουμε να πάμε γέρο στην Ολομέλη για να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό του Καναδά, τον κύριο Τρουντό. και αν ε, επιμένει η πλειοψηφία της ομάδας, μπορούμε να επανέλθουμε σε μεταγενέστερη τακτική μας συνεδρίαση και να συζητήσουμε το θέμα αυτό και πάλι. 28 Φεβρουαρίου, 12 το μεσημέρι, λίγη προθεσμία για τις τροπολογίες. 22 και 23 Μαρτίου θα εξετάσουμε τις τροπολογίες. Η έγκριση στην Επιτροπή Απασχόλησης ελπίζουμε να γίνει 12 και 13 Ιουλίου. Αν όλα πάνε καλά. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Καλή σας ημέρα.